Αγαπητοί συνάδελφοι, και τώρα να κάνουμε ψηφοφορία. Παρακαλώ καθίστε και ετοιμαστείτε για την ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία. Αφορά την έκθεση Σικία.